Έχουμε σήμερα την προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν για την κατάργηση του γυναικείου σεξουαλικού ακροτηριασμού και θα δώσω πρώτα πρώτα το λόγο στην κυρία Ζουμπέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η... Ο ακροτηριασμός των γενικών γενετικών οργάνων κοριτσιών και γυναικών είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Είναι πολλές ε, είναι εκατομμύρια γυναίκες που ε, γνώρισαν αυτή την οικογενειακή βία ε, σε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία στις δέκα μάλιστα έχει υποχρεωθεί σε υποχρεωτική σεξουαλική πράξη. Είναι ένας από τους χειρότερους, μια από τις χειρότερες μορφές βίας η παρέμβαση αυτή στη γυναικεία φύση. Η μορφή αυτή βίας κατά κοριτσιών σε νηπιακή ηλικία προκαλεί προβλήματα υγείας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Γυναικών ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει συγκεκριμένε δράσει ώστε να πάυσει αυτή η μορφή βία των ανδρών κατά των κοριτσιών και γυναικών. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική κατά τη βία που πλήττει τι γυναίκε, συμπεριλαμβάνοντα τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων. Όσοι έχουμε κάνει ω τώρα δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώ το φαινόμενο αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Γυναικών ε, για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που θεωρεί ότι μια συνολική στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν ένα σημαντικό βήμα. Δεν μπορεί πάντοτε τα δικαιώματα των γυναικών να μένουν ε, μια δεύτερη προτεραιότητα και να μην ε, λαμβάνουν την προσοχή που αξίζουν η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, Σύμβαση της ε, Ισταμπούλ, της Κωνσταντινούπολης, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας, θα πρέπει να προ... προβλέπει μάλλον ελάχιστους ε, κανόνες για τα δικαιώματα και την προστασία όλων των γυναικών και κοριτσιών. Αυτό είναι ένα βήμα που κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνει για να προστατεύσει τις γυναίκες και τα κορίτσια κατά τον ακροτηριασμό των γυναικείων οργάνων και άλλες μορφές βίας. Υπάρχει μια σειρά από διεθνή όργανα τα οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη να πάυσει η βία κατά των γυναικών και ο ακατηριασμό των γυναικείων οργάνων. Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η, ε, σύμβαση για την, ε, η δήλωση μάλλον για την η Σύμβαση για την Προστασία όλων των Δικαιωμάτων των Γυναικών και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Τα κείμενα αυτά και όσα προκύπτουν από αυτά είναι, σημαντικό και, είναι σημαντικά και πρέπει να εφαρμοστούν. Ο κριτηριασμό των ε, γυναικείων οργάνων αφορά πάνω από 140 ε, εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο. Τρία εκατομμύρια ε, κορίτσια, νήπια, κινδυνεύουν να γνωρίσουν αυτή τη μορφή βίας. Από το 2015 αρχίζουμε να μιλάμε για, νέες, για νέα δικαιώματα στην αυγή της νέας χιλιετίας. Θα πρέπει λοιπόν τα δικαιώματα των γυναικών να αποτελέσουν προτεραιότητα μεταξύ των νέων στόχων της χιλιετίας. Η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών θα πρέπει να θεωρηθεί ένας από τους πρωταρχικούς μας στόχους. Είναι σημαντικό να ορίσουμε συγκεκριμένους στόχους με συγκεκριμένα μέτρα και ε, πολιτικές συμφωνίες ώστε να αποφύγουμε τον ακριτηριασμό των γυναικείων οργάνων, να πετύχουμε την μείωση της παιδικής θνησιμότητας καθώς πρέπει να βελτιωθεί και η κατάσταση υγείας των ε, μητέρων και να προωθήσουμε τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κατηριασμός των γυναικείων οργάνων έχει τεράστιο αντίκτυπο στο αναπαραγωγικό κεφάλαιο και τη σεξουαλική υγεία των γυναικών. Το να πάψουν όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του εκτοτηριασμού των γυναικείων οργάνων, θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα που ε, ειδικό ε, στην περίοδο κρίσης που διανύουμε θα πρέπει να προσεχθεί. Ε, θα πρέπει οι περικοπές στα επιδόματα και την κοινωνική προστασία να πάψουν διότι έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κατάσταση των γυναικών. Όσες φροντίζουν ηλικιωμένες ενίοτε ή όσες εργάζονται σε συνθήκες επισφαλής. Θα πρέπει λοιπόν ήδη από σήμερα να προβλέψουμε μία συμπεριφορά που να μην στιγματίζει τις γυναίκες αυτές, να αποκλείει τη διακριτική συμπεριφορά, γιατί μπορεί να έχουν πέσει θύματα τέτοιου είδους ακροτεριασμού. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ποινές για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά να προλαμβάνουμε κιόλας για να ενημερώνουμε σωστά τι κοινότητε που πολλέ φορέ διαπράττουν τέτοιου είδου εγκλήματα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών. Και εδώ, ε, σε ένα πολιτικό σώμα, έχουμε το δικαίωμα τη πρωτοβουλία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε συντονισμένε στρατηγικέ για να πάψουν όλε οι μορφέ βία κατά των γυναικών, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των, ανθρώπων που συμπεριλαμβάνουν και αυτά των γυναικών και να καταπολεμήσουμε όλων των ειδών τι εγκληματικέ πράξει. Αυτό εφόσον θέλουμε να οδεύσουμε προς την κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Ζούμπερ. Ο Επίτροπος Φίλε. Σας κατευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Σήμερα είναι η Εθνή ημέρα κατά του γυναικείου σεξουαλικού ακροτηριασμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω, καταδικάζει τέτοιες τρομακτικές πρακτικές και έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τις γυναίκες και τα κορίτσια τέτοια φαινόμενα και στην Ένωση και εκτός αυτής όμως. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου να συζητήσει το θέμα. Ο σεξουαλικός ακροτηριασμός των γυναικών είναι μία βία έκφραση της ε, άνησης μεταχείρισης των φύλων και παραβίαση κατάφορη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε αναλόγως. Η Κομισιόν και η Ένωση στο σύνολό τη είναι διατεθειμένες και αποφασισμένες να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών μέσα στο έδαφος της Ένωσης αλλά και μέσω των εξωτερικών μας σχέσεων. Αυτό φαίνεται από το σχέδιο δράσης της Κομισιόν που εφαρμόζει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, την χάρτα των γυναικών και τη στρατηγική της Κομισιόν για την ισότητα των φύλων. Η Κομισιόν προσπαθεί να βελτιώσει τη συλλογή στοιχείων για αυτά τα φαινόμενα και να αυξήσει την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών τη χρηματοδότηση σε μήκη και όμικρον που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Το πιο πρόσφατη ένδειξη για τη δράση αυτή φάνηκε και στις 25 Νοεμβρίου πέρυσι από την σχετική μας δήλωση. Υπάρχει και θέμα κομεταχείρισης παιδών, γυναικών κοριτσιών δηλαδή που μπορεί να έχουν υποστεί κλειτοριδεκτομή. Το Κοινοβούλιο ζητάει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και στρατηγική για την καταπολέμηση αυτής της μορφής βίας κατά των γυναικών. Θα ήθελα να τονίσω ότι σε όλες τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν και τα μέτρα και τα μέτρα είναι συμπληρωματικά το ένα με το άλλο και αποτελούν στο σύνολό τους ένα πλαίσιο συνεπές με απτά αποτελέσματα και πλήρη χρήση των δικαιοδοσιών που έχει η Ένωση για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να εξαλείψουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών περαιτέρω. Ο σεξουαλικός ακροτηριασμός είναι συγκεκριμένη μορφή βίας που συχνά εφαρμόζεται με την πεποίθηση ότι θα κάνει καλό στο κορίτσι. Είναι βασικό να λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία του προβλήματος και γι' αυτό η Κομισιόν εφαρμόζει το σχέδιο δράσης αυτό για τον σεξουαλικό ακροτηριασμό μετά από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2012. Ας μιλήσω τώρα για το θέμα της νομοθετικής μας δράσης. Εδώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος με προτάσεις υπέρ των γυναικών και κατά της βίας κατά αυτών όπως η οδηγία για το δουλεμπόριο κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της παιδικής πορνογραφίας και αυτά συμπληρώνονται και με κανονισμό που εφαρμόζεται και σε αστικά θέματα. Όλα αυτά τα νομοθετήματα τονίζουν την ανάγκη για συγκεκριμένη και κατάλληλη αναλογική προστασία από τη βία κατά των γυναικών. Έχουμε το απαραίτητο πλαίσιο για να προστατεύσουμε τις γυναίκες κατά όλων των μορφών βίας αλλά αυτά πρέπει και να εφαρμοστούν αποτελεσματικά από τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Η Κομισιόν βοηθάει τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό και θα υποπτεύσει και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Εκτός αυτών υπάρχουν και μέτρα μη νομοθετικά για πληροφόρηση, για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και χρηματοδότηση. Αυτά τα μέτρα ήδη συμβάλλουν στην στήριξη των χωρών μελών για την πρόληψη της βίας. Για τι εξωτερικέ σχέσει σα υπενθυμίζω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία είναι αναπόσπαστο τμήμα όλης μας της πολιτικής για κάθε πρόγραμμα στήριξης κάποιας χώρας και τα δικαιώματα των γυναικών και κοριτσιών συμπεριλαμβάνονται φυσικά. Αρχίζουμε επίσης τώρα να εφαρμόζουμε μία προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα με την οποία αναγνωρίζουμε τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ως ε, νόμιμους εταίρους και συνομιλητές μας. <coughs> Έχουμε συμμετάσχει ενεργά και σε διεθνείς πρωτοβουλίες προώθησης όλων αυτών των θεμάτων. Συστηματικά θέτουμε το θέμα του σεξουαλικού ακροτηριασμού στους διαλόγους μας με αφρικανικές ε, χώρες, χώρες του Ειρηνικού και της Ασίας και θέλουμε να διασφαλιστεί ότι ο σεξουαλικός ακροτηριασμός θα απαγορευτεί. Επίσης στηρίζουμε προσπάθειες lobbying για την προώθηση των γυναικείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το capacity building καθώς και την πληροφόρηση για όλους, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας ετοιμάζουμε και μια περιφερειακή καμπάνια για τον σεξουαλικό ακροτηριασμό που θα την εφαρμόσουμε και σε αντιπροσωπείες μας σε τρίτες χώρες το 2014. Επίσης χρηματοδοτούμε προγράμματα από 6 με 12, την περίοδο 6 με 12, 17 προγράμματα στήριξης ε, της καταπολέμησης του σεξουαλικού ακροτηριασμού για, ε, σε ύψος περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ προγράμματα της UNICEF ας πούμε για το σεξουαλικό ακροτηριασμό στην Αίγυπτο, Σουδάν, Ερυθρέα και αλλού. Ο εκδημοκρατισμός, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέματα που στήριξε η Ένωση σε πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σας κατευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Φίλε. Ακολουθούν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Πρώτη κυρία Γκάμπριελ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. καταρχά χαίρομαι που ψηφίζουμε σήμερα το ψήφισμα αυτό και την προφορική ερώτηση για την εξάλληψη του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ομόφωνα εγκρίθηκε στην Επιτροπή ελπίζω και στην Ολομέλεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράξει αυτή την ευκαιρία για να στείλει ένα σαφέ μήνυμα ότι είναι προσιλωμένο στην προσπάθεια αυτή να τερματιστεί αυτή η κατάφορη και ομή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι θα συνάδουμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα την κυρία Ρέντινγκ που ε, ξεκίνησε αυτή την εκστρατεία για μηδενική ανοχή, άρχισε τη συζήτηση και ευαισθητοποίησε τον κόσμο σε αυτή τη μάστεγα. Επιτρέψτε μου να επιμείνω σε μερικά σημεία που θεωρώ σημαντικά για την εξάλληψη που έχουμε ως στόχο. Πρώτον, ο ακροτηριασμός των γυναικείων ε, γεννητικών οργάνων συνιστά κατάφορη και ε, αδιαφυσβήτητη παραβίαση των δικαιωμάτων, ε, επέμβαση στον ψυχισμό και στο σώμα και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία που να ισχύει παράδοση, θρησκεία, πολιτισμός Επίσης θυμίζω ότι συμβαίνει και στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες με τις οποίες έχουμε σχέσεις και δεν μπορούμε αυθαίρετα και ε, συνολικά να στιγματίζουμε την Αφρικανική Ήπειρο γιατί διαφέρουν ε, οι πραγματικότητες από χώρα σε χώρα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ολοκληρωμένη και γενική στρατηγική για να υπάρχει και μία συνέπεια ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική και να μην αρκούμαστε να δίνουμε μαθήματα στους άλλους για το θέμα αυτό. Εξαρτήσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης χρειάζονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, επιμένω, θα πρέπει και οι άνδρες και τα γόρια να συμμετάσχουν σε αυτή την εξαρτία συνειδητοποίησης. Αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να εξαλειφθεί διάλογο στο εσωτερικό μιας κοινότητας είναι πάρα πολύ κρίσιμος για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο στόχο μας. Και τέλος, δεν θα πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ε, της ε, σε ιατρικό περιβάλλον ε, που χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Ακροτηριασμός είναι και αν γίνει σε στήρο περιβάλλον από γιατρό αλλάζει. Κυρίε και κύριοι, Επίτροπε, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τη μηδενική ανοχή για το φαινόμενο αυτό. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία εγώ και να απευθυνθώ στη διεθνή κοινότητα, όχι μόνο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να τερματιστεί αυτή η μάστιγα, επαναλαμβάνω. Και ευχαριστώ τους αραλέους εκείνους άνδρες και γυναίκες που καθημερινά αγωνίζονται σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ κυρία Στρέλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ήδη υπόθηκε. Είναι περίπου 140 εκατομμύρια οι γυναίκες που ήδη έχουν υποβληθεί στον εκατηριασμό των ε, γενετικών τους οργάνων. Ε, κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια κορίτσια και έφηβες ε, πέφτουν θύματα εκατηριασμού. Είναι μία κάθε έξι λεπτά Πολλές φορές αυτή, αυτός ο κατηριασμός γινόταν περίπου στην ηλικία των 8-9 ετών. Αυτή τη στιγμή ε, τα κοριτσάκια αυτά μπορεί να είναι 2 ή 3 ετών. Αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα σε τρίτες χώρες, σε πολλές τρίτες χώρες. Όμως παρατηρείται και σε συγκεκριμένες κοινότητες οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 98% ε, των ε, γυναικών και κοριτσιών ακροτηριάζονται σε τηλετουργικά που συμμετέχει η οικογένεια ε, των θυμάτων και αυτό είναι μια γιορτή στο Μαλί. Ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων λοιπόν πολλές φορές είτε συμβαίνει στις χώρες προέλευσης είτε στην Ευρώπη είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μάστιγα και πρόκειται για μια πραγματικά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ε, συμπεριφέρονται με συγκατάβαση και αδιαφορία σε τέτοιου είδους εγκληματικές ε, δράσεις με πρόσχημα την παράδοση που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ψυχολογική και σωματική υγεία των γυναικών. Οι έφηβες γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε ακροτηριασμό ε, αντιμετωπίζουν πολλές σοβαρές συνέπειες, θάνατο από αιμορραγία ή από μόλυνση ή πιο εύκολη μετάδοση ασθενειών όπως ο τέτανος και η πατήτιδα ή ε, σεξουαλικές, σεξουαλικώς ασθένειες ή περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του τοκετού. Ε, οι ψυχολογικές συνέπειες επίσης είναι πολύ σοβαρές και για αυτό το λόγο τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να προβλέψουν ε, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και ψυχολογικής στήριξης, καθώς και ενημέρωση για τα θέματα αναπαραγωγικής σεξουαλικής υγείας, ώστε να προστατεύονται τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα τέτοιου είδου βία. Έχουμε πολλά που πρέπει να κάνουμε και έχουμε υποχρέωση να κάνουμε περισσότερα για αυτέ τι νέε, για αυτέ τι έφηβε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Στρέλα και κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το 2004 θεσπίστηκε η σημερινή Παγκόσμια ημέρα μηδενική ανοχή των ακροτών των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Έκτοτε έχουν γίνει πολλά, αλλά πολύ λίγα παραμένουν αυτά. Παγκοσμίω πρόκειται για πάνω από 140 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια. Είναι ομοί και βία. Στην Αυστρία ε, υπάρχει η πλατφόρμα stopfgm.net που κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν, να ενημερώσουν και τελικά να καταγγείλουν ε, αυτή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το τελειτουργικό που αποβαίνει που συχνά και μοιραίο. Πολλοί κάνουν πολλά και πολλά κράτη και πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με το θέμα αυτό και με πολύ μεγάλη δέσμευση. Ε, όσο παραμένουν αυτές οι πρακτικές όμως του ακροτηριασμού είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θα πρέπει να έχουμε μια ενιαία στρατηγική τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και ελπίζω να μπορέσουμε να τερματίσουμε και να εξαλείψουμε αυτό το τελετουργικό επαναλαμβάνω και να είμαστε ομόφωνοι απέναντι σε τρίτες χώρες για να το διατρανώσουμε αυτό. Μηδενική ανοχή και τίποτα άλλο αλλά δεν επιτρέπεται με ευρωπαϊκά κονδύλια να υποστηρίζονται τρίτες χώρες όπου αυτή η πρακτική ε, παραμένει αποδεκτή κοινωνικά. Τέλος, διερωτώμε σε ποιο κόσμο ζούμε εάν δεχόμαστε γυναίκες και κορίτσια να υφίστανται αυτή τη βία. Και θέλω να πω ότι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που σιάζει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Ρωμέβα για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Το Δεκέμβριο του... Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν στη Γενική Συνέλευση ένα ψήφισμα ε, το οποίο καλεί ε, να δημιουργηθεί μια στρατηγική ε, προς την εξάλληψη αυτού του φαινομένου. Στην Ευρώπη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπολογίζει ότι 500.000 γυναίκες ζουν με τις συνέπειες ε, αυτού που είναι σαν το πληθυσμό της Μάλτας και κάθε χρόνο κινδυνεύουν 180.000 γυναίκες. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει το ρόλο της για να τερματιστεί αυτή η πρακτική. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστά στοιχείο κλειδί ε, για την απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών της Γενικής Συνέλευσης. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Χρειάζεται μια διακλαδική, διεπιστημονική προσέγγιση. Ε, επιμένουμε στην ανάγκη των προληπτικών δράσεων. Τι σημαίνει αυτό να εργαζόμαστε με τις κοινότητες αυτές και για τις κοινότητες αυτές με νέους και νέες. Σημαίνει ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα σχετικά με το φύλλο και να ε, σταματήσει σε κάθε κοινότητα αυτό. Πρόληψη σημαίνει επίσης και κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματιών που πρόκειται να συναντήσουν γυναίκες και κορίτσια. Ε, αλλά δεν σημαίνει δίωξη η πρόληψη. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την ποινικοποίηση. Δεν υπάρχει καθόλου, καμία ένδειξη σήμερα ότι η καταστολή ε, απαλήφει το φαινόμενο. Χρειάζονται μέτρα προστασίας των παιδιών και να καταλάβουμε ότι ε, αυτή η πρακτική αφορά όλη την κοινωνία. Οι φυλακές, ε, οι διώξεις ε, η απομάκρυση των γονέων από το παιδί μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να συγχαίουμε την πρόληψη με την καταστολή, την κατανόηση με το φόβο. Αυτό που χρειάζεται είναι να αλλάξει το σύστημα αυτών των πεπιθήσεων ε, και ε, η πρακτική να τερματιστεί. Είναι ένας αγώνας δρόμου, αγώνας αντοχής που χρειάζεται στοιχεία ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον επιπολασμό, για να ξέρουμε ε, τι ισχύει και ποιες είναι οι σωστές απαντήσεις και οι πολιτικές. Εμείς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να υποστηρίξουμε όσους εργάζονται ήδη προς την κατεύθυνση αυτή και χαίρομαι πάρα πολύ που το ψήφισμα ε, υποστηρίζει αυτούς στην Ευρώπη. Εμείς που θα είμαστε ξανά υποψήφοι για την επόμενη θητεία Θέλουμε να δείξουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια υπογράφοντας την υπόσχεση ότι ε, θα τερματιστεί. Αυτό υπάρχει μια σχετική πλατφόρμα που κυκλοφορεί. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Κουδάκη, Παρακαλώ. Thank you. Ο ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων είναι μια αποτρόπαιη και ε, βάρβαρη πράξη που διαπράτεται κατά των νεαρών κοριτσιών γυναικών. Ξέρουμε σήμερα ότι περίπου 500.000 κορίτσια στην ηλικία των τριών βρισκόνται σε κίνδυνο στην Ευρώπη. Στον Ηνωμένο Βασίλειο μόνον εκτιμούμε περίπου σε 65.000 τα ε, αριθμό των κοριτσιών που κινδυνεύουν. Οι περισσότερε ζουν στην εκλογική μου περιφέρεια, το Λονδίνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η μορφή αυτή ακροτηριασμού ε, θεωρήθηκε έγκλημα το 1995, όμως τα τελευταία 19 χρόνια δεν υπήρξε ούτε μία δίωξη, ούτε μία υπόθεση δίωξης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινήσαμε τον αγώνα για να σταματήσει αυτή η βάρβαρη ε, παράδοση και η πρώτη λονδρέζικη εφημερίδα, London Evening Standard, βρέθηκε στην ε, πρώτη γραμμή του αγώνα αυτού, ε, υπογραμμίζοντας το φαινόμενο, ενημερώνοντας το κοινό για την πρακτική αυτή και δεν καταφέραμε να πάυσει το φαινόμενο αυτό. Παρακαλώ του υπόλοιπου ευρωβουλευτέ να ενώσουν τι δυνάμει του μαζί μου για την καταπολέμηση αυτή τη κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Σήμερα, Διεθνή ημέρα για την μηδενική ανοχή κατά του ακροτηρισμού των γυναικείων γενετικών οργάνων, αλλά και κάθε ημέρα. Γι' αυτό υποβάλαμε αυτό το ψήφισμα ω ένα πρώτο βήμα για να πάυσει ο ακροτηρισμό των γυναικείων γενετικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την επόμενη εβδομάδα θα διοργανωθεί μια ακρόαση όπου θα προεδρεύω για το θέμα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο με παρουσίαση πολλών δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου να εξαλειφθεί αυτή η πρακτική σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι θα γίνει σύντομα και δημόσια κρόαση και στη δική μου εκλογική περιφέρεια στο Λονδίνο με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων ε, για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και είσαστε όλοι ευπρόσδεκτοι στι εκδηλώσει αυτέ. Πρέπει σε όλα τα κράτη-μέλη να προωθηθεί μια τέτοια πολιτική μηδενική ανοχή. Πρέπει να στηρίξουμε τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που σε όλο τον κόσμο εργάζονται για να εκπαιδεύσουν, να ενημερώσουν τι ε, κοινότητε όπου αυτά συμβαίνουν, να καταλάβουν ότι αυτή είναι μια παράδεκτη πρακτική και μιλάμε για ε, πραγματική βία κατά των παιδιών που δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Το ψήφισμα αυτή τη εβδομάδα είναι μια έκκληση να αναλυθεί δράση. Σήμερα σα ζητώ να ενώσετε τι δυνάμει σα μαζί μου για να υπάρξει τέτοιου είδου δράση. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κυρία Γιανακουδάκη. Η κυρία Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα 6 Φεβρουαρίου είναι η δέκατη επέτειος της θέσπισης της ημέρας για μηδενική ανοχή στον ακριοτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Πάνω από 3.000 γυναίκες στην Ιρλανδία έχουν πέσει θύμα αυτής της πρακτικής σύμφωνα με υπολογισμούς παρά το γεγονός ότι ε, απαγορεύεται από τον νόμο και ε, χιλιάδες κορίτσια και γυναίκες κινδυνεύουν σε όλη την Ευρώπη να υποστούν έστω και παράνομα αυτή την πρακτική ή ε, τους πηγαίνουν πίσω στις χώρες προέλευσης των γονιών τους. Αυτό αναμφίβολα είναι μια πρακτική βάρβαρη και αρχαϊκή που θα πρέπει να σταματήσει πολλές γυναίκες που υποχρεώνται να την υποστούν πεθαίνουν από αιμορραγία ή από λοιμώξεις γιατί είναι βρώμικα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Εδώ πρόκειται για μια επέμβαση στη φυσιολογία, στη φυσιολογική ζωή και στο σώμα τους ε, γιών κοριτσιών και ε, υγιή γεννητικά όργανα ακροτηριάζονται. Είναι πολύ μεγάλος ο πόνος και τεράστιες οι συνέπειες και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Μέχρι και στον τοκετό υπάρχουν δυσκολίες και μπορεί να προκληθεί και βλάβη στο νεογέννητο. Οι γυναίκες που επιζούν ε, αντιμετωπίζουν το φόβο και μακροπρόθεσμες συνέπειες της λίμωξης. Υπάρχει ε, το Εθνικό Δίκτυο Μεταναστριών που ζουν στην Ιρλανδία και έχουν κάνει σπουδαία δουλειά εδώ, αλλά λυπάμαι που είναι περιορισμένη η εμβέλειά του. Το γεγονός ότι το συζητούμε και σήμερα σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει αρκετά. Στην ίδια μου την εκλογική περιφέρεια, στη Βόρεια Ιρλανδία, ενημερώνονται ε, οι δάσκαλοι όταν βλέπουν κορίτσια να απουσιάζουν ε, ε, πολύ καιρό από το σχολείο, πηγαίνουν και επισκέφτονται τις οικογένειές τους από το φόβο μήπως έχει γίνει ακροτηριασμός. Είναι παράνομο αυτό στην Ιρλανδία, αλλά πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να συνειδητοποιήσει ο κόσμος στον ακροτηριασμό αυτό. Διεθνώς αναγνωρίζεται ως παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών και κοριτσιών και αντανακλά μια βαθιά ριζωμένη αδικία μεταξύ και ανισότητα μεταξύ των φίλων και βαριά μορφή διάκρισης κατά των γυναικών. Σχεδόν πάντα γίνεται σε ανήλικες και παραβιάζει και τα δικαιώματα των παιδιών διαδοχικές προεδρίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου απέτυχαν να το καταστήσουν προτεραιότητα. Και είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Χαίρομαι που η Γενική Συνέλευση ε, του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 2012 ενέκρινε ένα ψήφισμα για την εξάλληψη αυτού του ακροτηριασμού και το καλωσορίζω, επαναλαμβάνω ότι σήμερα το συζητούμε αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ήδη έχει εγκρίνει ένα σχετικό ψήφισμα αλλά χρειάζονται πολύ πολύ περισσότερα ακόμα να γίνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μοργκάντη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα δεδομένα που διαθέτουμε για αυτή την φρικτή πρακτική ε, πραγματικά εντυπωσιάζουν. Ε, ακόμη και αν δούμε τι έχει συμβεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 25.000 γυναίκες τουλάχιστον στην Ήπειρό μας που έχουν πληγεί από αυτό το φαινόμενο. Είναι 125 εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο βέβαια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο σοβαρά τα γεγονότα που αφορούν την ε, δική μας Ήπειρο. Μιλάμε για νοοτροπίες και πολιτισμού πολύ μακρινούς από τους δικούς μας. Όμως σήμερα τον 21ο αιώνα είναι πραγματικά τρομακτικό να πρέπει να μιλάμε για τέτοια ε, δεδομένα. Σήμερα βάσει του παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα των γυναικών στην Ιταλία έχουμε περίπου 35.000 γυναίκες που ε, έχουν πληγεί από τέτοιου είδους πρακτική και είναι μισό εκατομμύριο αυτές που κινδυνεύουν. Πρέπει αμέσω να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και πρέπει να υπάρξουν σοβαρέ ποινέ για όσου διαπράττουν αυτό το είδου τα εγκλήματα. Διότι είναι απαράδεκτο στην Ιταλία και στην Ευρώπη να διαδίδεται τέτοια βαρβαρότητα. Θα πρέπει ε, να ε, αυτή η παράλογη, επικίνδυνη και χωρί νόημα πρακτική να αντιμετωπιστεί σαν εκδήλωση μια υποκουλτούρα με θρησκευτικά προσχήματα. Σήμερα, τη Διεθνή ημέρα για το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει να έχουμε την τόλμη να πούμε τα πράγματα ανοιχτά, να ορίσουμε από πού προέρχεται αυτή η πρακτική, από ποιες χώρες, ποιες είναι οι θρησκείες που την ανέχονται, ε, ξεκινώντας από το Ισλάμ και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν φτάνει μόνο μια ευρωπαϊκή συνολική στρατηγική κατά της ε, βίας ε, λόγω φύλου που μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Είναι συγκεκριμένη πολιτιστική χώροι όπου αυτά καλλιεργούνται. Στην Ευρώπη λοιπόν που θέλουμε να προασπιστούμε την χριστιανική μας ε, θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι είμαστε διαφορετικοί να μην έχουμε ανοχή για αυτούς που λένε ότι είναι διαφορετικοί από εμά με, με τέτοιο θράσος. Διότι μπορεί να βρίσκουν πολλές δικαιολογίες για να διαπράττουν τέτοιες απετρόπες πρακτικές που προκαλούν μακροπρόθεσμα ε, τέτοιο πόνο. Σας ευχαριστούμε κύριε Μοργκάντη και τώρα η κυρία Χιμένες Μπεθερίλ Μπαριγιό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα επαναλάβω τον ορισμό του ακροτηριασμού των γενικών γενετικών οργάνων. Της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας είναι. Είναι επίγον να μπει φρένο σε αυτή την ε, οδύνη σε αυτά τα δεινά των γυναικών. Είναι η ολική ή η μερικη κλειτοριδεκτομή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. 140 εκατομμύρια κοριτσιών και γυναικών υπέστησαν αυτού του είδους τη βία σε όλο τον κόσμο που στιγματίζει τα κορίτσια στην παιδική του ηλικία και στην εφηβεία. Αυτή η ομή και βία πρακτική δεν γίνεται μόνο σε τρίτες χώρες αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, φτάνει στον εισηγητικό αριθμό που ακούσαμε, 500.000 και ακόμα πολλές περισσότερες που ε, έπονται. Γνωρίζουμε ότι ο ακροτηριασμός αυτός γίνεται σε εκτρές συνθήκες υγιεινής και πολλές φορές είναι ανεπανόρθωτες οι συνέπειες για την υγεία του κοριτσιού. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι κατοχυρωμένη σε νόμους και στις χώρες μας και διεθνώς και μας υποχρεώνει αυτό να μην ανεχόμαστε αυτή την πρακτική. Δεν στέκει καμιά δικαιολογία και καμιά πολιτιστική παράδοση. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε εγκρίνει διάφορα ψηφίσματα προς την κατεύθυνση κατεύθυνση της καταπολέμησης, στην οδηγία για την προστασία ε, των δικαιωμάτων των θυμάτων που ήμουν εισηγήτρια ε, ζήτησα να τιμωρείται αυτό και στα 28 κράτη-μέλη. Η χώρα μου, η Ισπανία, έχει ειδική ποινική νομοθεσία, αλλά δεν υπάρχει ομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε κοινή προσέγγιση με κοινά στοιχεία και ανταλλαγή δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα πρέπει να λάβει στεναρή θέση απέναντι σε τρίτε χώρε που δεν καταδικάζουν αυτού του είδου τη βία κατά των γυναικών. Είναι πολλά τα θύματα που δεν έχουν φωνή, που δεν ακούγονται και είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε τη δική μας φωνή για να εξαλειφθεί αυτή η βία κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 21ο αιώνα κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σενεζίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο, γυναικείος, ο ακροτηριασμός των γυναικείων γενετικών οργάνων είναι μια απαράδεκτη μορφή ε, βίας ε, η οποία ε, αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως ε, αλλάζει την ταυτότητα της γυναίκας του νεαρού κοριτσιού. Αφορά 500.000 ε, γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, αλλά σίγουρα τα δεδομένα αυτά υποτιμούν τον αριθμό των γυναικών που πρέπει να κινδυνεύουν στην πραγματικότητα στα κρατη μέλη. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει τι έχει γίνει ως τώρα για την καταπολέμηση του ακροτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός αυτής όμως θα πρέπει τέτοιου είδου δράσει να αποτελέσουν μέρο μια συνολικότερη στρατηγικής, ώστε να υπάρξει νομοθεσία που να προστατεύει πραγματικά τι γυναίκε από τον ακροτηριασμό των ε, γυναικείων γεννητικών οργάνων. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με τι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρούν εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωκοινοβούλιο θέλει ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει την ε, παράταση λειτουργία των οργάνων που τη συνεργασία των κρατών μελών θέματα αυτά με, για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών συμπεριλαμβανόμενης ε, της μορφής αυτής βίας. Για τα δεδομένα εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και για τη δράση μα εκεί και πάλι χρειάζεται πολλή δουλειά. Χρειάζονται διορθωμένες πολιτικές ώστε οι χώρες που έχουν στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρνούνται να αναλάβουν δράση κατά του φαινομένου αυτού να κάνουν επιτέλους κάτι. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει μια ρήτρα που να καλύπτει τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων στι διαπραγματεύσει τη, προκειμένου να επιτύχει συμφωνίε με τέτοιου είδου χώρε. Τι γίνεται ω προ αυτό. Έχουμε το καθήκον να προστατεύσουμε τα θύματα ε, αυτή τη μορφή βία. Και ω προ την πρόληψη θα πρέπει να προσβλέψουμε ψυχολογική στήριξη για του ανθρώπου αυτού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόκειται για μια μορφή βασανισμού των γυναικών και δεν είναι κάτι που συμβαίνει μακριά από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θέλουμε να φανταζόμαστε, αλλά δεν ισχύει αυτό. Μισό εκατομμύριο γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θύματα αυτής της πρακτικής και 125 εκατομμύρια είναι θύματα σε όλο τον κόσμο. Το να είναι κανεί θύμα τέτοιου είδους ακροτηριασμού είναι πραγματικά σαν να είναι, θέμα, ε, σαν να είναι θύμα σοβαρότατων ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου που κανονικά έπρεπε να προστατεύονται στην εποχή μας και όλα ε, όσα έχουμε επιτύχει να προστατεύσουμε έχουμε, έχουν καταρρεύσει εάν αυτό δεν το έχουμε πετύχει. Με την έκθεση Εστρέλα πρόσφατα μιλήσαμε για την προστασία των γυναικών. είδαμε πόση προσοχή έλαβε το θέμα αυτό, πόσο, τραβά, πόσο προσελκύει την προσοχή των πολιτών τέτοια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Λάβαμε τόσα mail για τα θέματα αυτά. Η υγεία λοιπόν, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των γυναικών είναι κάτι που αφορά όλους. Είναι πολύ περίεργο να μην γίνεται τίποτα για το φαινόμενο αυτό. Μιλάμε για μια μορφή βασανιστηρίου, ε, για σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες που μπορεί να κρατήσουν μια ολόκληρη ζωή. Δεν γίνονται αρκετά λοιπόν ε, σε κάποιες χώρες για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, αλλά πρώτα να κοιτάξουμε τι γίνεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισό εκατομμύριο γυναίκες είναι τεράστιος αριθμός για τη δική μας την Ήπειρο. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε τις υπόλοιπες χώρες μόνο και να μην βλέπουμε τι γίνεται στο σπίτι μας. Ε, καλωσορίζουμε λοιπόν το σχέδιο δράσης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που αντιμετωπίζει και το φαινόμενο αυτό, αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερο και στον πέδο της πρόληψης. Ευχαριστούμε κυρία Μακλάρκιν για δύο λεπτά. Πριν από δύο χρόνια Είχα μιλήσει για την περίπτωση του Άρες Ντιούι που τώρα είναι πρεσβευτής για την κατάργηση του γυναικείου σεξουαλικού ακροτηριασμού. Έχω ξαναπεί ότι η περίπτωση εκείνη με είχε συγκινήσει μέχρι δακρύων. Η τρομακτική αυτή πρακτική εφαρμόζεται σε εκατομμύρια παγκοσμίως. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πρακτικής αυτής και γι' αυτό είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ να ζητήσουμε από την Κομισιό να εφαρμόσει τις συστάσεις της για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να καταργήσουν αυτή τη βάρβαρη πρακτική που αφορά τόσα εκατομμύρια και μέσα στην Ένωση ακόμα. Πρέπει να καταλάβουν οι γυναίκες ότι η πρακτική αυτή είναι τεράστια βιοπραγία εναντίον τους και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και τα κράτη-μέλη τα ίδια θα κατανοήσουν καλύτερα πόσο διαδεδομένη είναι η πρακτική αυτή για να προβλέψουν τις κατάλληλες κυρώσεις. Επίσης πρέπει η Κομισιόν να δει και στις τρίτες χώρες πώς μπορεί να καταργηθεί η πρακτική αυτή. 125 εκατομμύρια γυναίκες ενδιαφέρει. Και είναι πρόβλημα και υγείας. Η πρακτική αυτή πρέπει να καταδικαστεί παγκοσμίως και υποστηρίζω πλήρως τον Επίτροπο Φιούλε και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να κάνουν κάτι στις χώρες που δεν θα αντιδράσουν. Πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν να καταργηθεί αυτή η βάρβαρη πρακτική παγκοσμίω. Ευχαριστούμε κυρία Μακλάρκιν. Ο κύριος Μάρφης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς δεν βρίσκω εκπληκτικό αλλά ιδιαστικό ότι οι ακροδεξιοί ευρωβουλευτές όπως Μοργάνο προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν με την πρόφαση αυτής της βάρβαρης πρακτικής ένα επιχείρημα για να προωθήσουν ισλαμοφοβικά και ρατσιστικά προγράμματα και ιδέες οι αφρικανικοί πολιτισμοί που βασίζονται στο Ισλάμ δεν είναι οι μόνες που εφαρμόζουν αυτή τη βάρβαρη πρακτική. Δέστε τι βιοπραγίες κατά των γυναικών σημειώνονται μέσα στην Ένωση σε χριστιανικούς πληθυσμούς. Την οικιακή βία που πλήττει μία σε πέντε γυναίκες. Δεν είναι εδώ το θέμα να επιβληθούν μεγάλες ευρωπαϊκές αξίες σε άλλους πολιτισμούς. Το θέμα είναι ανθρωπίνων, γυναικείων, παιδικών δικαιωμάτων για δικαιώματα για τα οποία μάχονται και οι πληθυσμοί της Αφρικής και αλλού. Υπάρχει το μυθιστόρημα Possessing the Secrets of Joy που περιγράφει τα βάσανα που υποφέρουν οι γυναίκες από το γάμα σίγμα άλφα. και έρχομαι εδώ στο βασικό θέμα του γάμα σίγμα άλφα. είναι μία έκφραση καταπίεσης των γυναικών και τρόπος άρνησης του, της σεξουαλικής ταυτότητάς τους. Η Ένωση έχει εδώ ευθύνη. Κάθε χρόνο 20.000 γυναίκες υπολογίζεται ότι ζητούν άσυλο κατά τέτοιων πρακτικών στην Ένωση και πολλές ακόμη για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Οι μαρτυρίες από τα θύματα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει αρκετή γνώση για το θέμα και τόσο πολλές, αυτό το δείχνει το γεγονός ότι τόσο πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν στείλει πίσω τις γυναίκες αυτές στις χώρες από όπου προέρχονταν. Έχουν την υποχρέωση τα κράτη-μέλη να προστατεύσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια από το γάμα σίγμα α. Έχει βέβαια κηρυχθεί παράνομη σε μερικές χώρες, αλλά χρειάζονται περισσότερη ανάλογη νομοθεσία και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για να μειωθεί η εξάρτηση των γυναικών από παραδοσιακούς σε εισαγωγικά γιατρούς που εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μέρφυ. Πριν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κορατσαμπίλτ να υποδεχθώ εξ ονόματος όλων μας αρμενική αντιπροσωπεία που συμμετέχει στη 14η συνέλευση της κοινή ε, Συνέλευσης Συνεργασίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αρμενίας. Καλώς ήρθατε. Κυρίως καλώς ήρθατε εσείς κύριε Φαρμανιά που προεδρεύετε. Θα παρευρεθείτε σύντομα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ελπίζουμε συνεργασία